Καλημέρα σας. Α, μάλιστα μου απάντησε κάποιος και προχωρούμε στην ημερησία διάταξη. Σήμερα έχουμε τη μελέτη για τη μείωση της ε, αποχώρησης από τα σχολεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δούμε τι θα πει η κυρία Άννα Μαρία Νεβάλα από το Ενωμένο Βασίλειο. Κυρία Νεβάλα, η πέστε μας σας παρακαλώ. Πολύ σας ευχαριστώ. Θέλω ευχαριστήσω την πρόεδρο της Επιτροπής και τους συναδέλφους από την ε, από το Τμήμα Πολιτικής Β του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με προσκάλεσαν να παρουσιάσω τα πεπραγμένα μας του χειμώνα σε σχέση με την αποχώρηση από το σχολείο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα και νιώθω ιδιαίτερα έντονα για τα θέματα αυτά. Έχω εργαστεί πάρα πολύ καιρό για τα θέματα αυτά. Είναι μια μεγάλη τιμή για μένα που με έχετε φέρει εδώ. Λέγομαι Αννα Μαρία Αν Μαρή Ζω στην Αγγλία αλλά έρχομαι από τη Φιλανδία και εκπροσωπώ μια ομάδα από ερευνητές και ανθρώπους που ασχολούνται με τα θέματα της εκπαίδευσης που κάνουν αυτό το project που σας παρουσίασα, που σας είπα προηγουμένως, αυτό το χειμώνα. να σας πω λοιπόν καταρχήν ποιοι ήταν οι στόχοι μας, τι μας ζητήσανε να κάνουμε, τι προσπαθήσαμε να κάνουμε τους τελευταίους μήνες. Ο στόχος μας ήταν να δώσουμε συστάσεις για τους εμπλεκόμενους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, να εξηγήσουμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη σε σχέση με το θέμα αυτό και να δώσουμε παραδείγματα πολιτικών οι οποίες είναι ευστοχές αυτή τη στιγμή και επίσης μας ζητήσανε να συζητήσουμε κατά τη διάρκεια ενός τετραμήνου τον προηγούμενο χειμώνα και κοιτάξαμε τα κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται με τους νέους, με ενώσεις μαθητών, με ενώσεις και με ανθρώπους που εργάζονται με τα άτομα τα οποία έχουν αποχωρήσει πρόωρα από το σχολείο κτλ. Όπως σας είπα, εστιάσαμε σε εννέα χώρες από όλη την Ευρώπη, από τα ανατολικά ως τα δυτικά, από τα νότια ως τα βόρεια, με υψηλό επίπεδο αποχώρησης, χαμηλό επίπεδο αποχώρησης, με χώρες που μειώνεται αυτό το ποσοστό και με χώρες όπου αυξάνεται αυτό το ποσοστό. <clears throat> Φιλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λιθουανία, κάτω Πολωνία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Κυρίως το τμήμα της Αγγλίας μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ποιοι είμαστε τώρα. Εγώ έρχομαι από ένα ερευνητικό φορέα που περιλαμβάνει ερευνητές από άλλες 20 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. που προανέφεραν και φυσικά είχαμε διαφορετική προέλευση και διαφορετική πείρα. Όλοι μας ήμασταν ερευνητέ στον τομέα της ε, παιδείας, αλλά είχαμε και ακαδημαϊκούς και άτομα τα οποία λειτουργούν ως εκπαιδευτικοί καθημερινό επίπεδο ποια είναι τα εκπαιδευτικά προβλήματα σε σχέση με την πρόορη αποχώρηση από το σχολείο και είχαμε και ένα μέλος της ομάδας μας που είχε και εμπειρογνωμοσύνη στην ανάπτυξη πολιτικών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πρόορης αποχώρησης και μετά στην εφαρμογή τους. Πάω τώρα στη μελέτη και στις, στα κύρια συμπεράσματά μας. Είναι φανερό λοιπόν ότι το πρόβλημα της προώρησης αποχώρησης από το σχολείο είναι ένα πρόβλημα όχι μονάχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ... Για δύο κύριους λόγους είναι κύριο θέμα πολιτικής. Πρώτον γιατί μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των ατόμων που έχουν αποχωρήσει πρόωρα από το σχολείο και φυσικά λόγω και του γενικότερου κοινωνικού αντικτύπου. Υπάρχουν πολλά στοιχεία και στο εθνικό και στο, εθνικό και στο παγκόσμιο επίπεδο ότι αυτοί οι οποίοι αποχωρούν νωρίς από το σχολείο βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και κοινωνικά και οικονομικά σε σχέση με, τους, με τα άτομα της ίδιας ηλικιακή ομάδος. Και επομένω αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα για την κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Δεν σημαίνει αυτό για όλους. Υπάρχουν πολλοί νέοι οι οποίοι φεύγουν από το σχολικό σύστημα και μπορεί στη συνέχεια να έχουν μια επιτυχημένη καριέρα. <clears throat> Δυστυχώς όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο για την πλειοψηφία αυτών που αποχωρούν νωρί από το σχολείο. Κατά κύριο λόγο είναι άνεργοι βασίζονται σε κοινωνικά επιδόματα και βρίσκονται λοιπόν σε πολύ πιο δύσκολη θέση από τους ομολόγους τους που είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι. Επίσης έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες και έχουν και περισσότερα προβλήματα υγείας από το μέσο πληθυσμό. Αυτό σημαίνει ότι η αποχώρηση, η πρόορη αποχώρηση σαν κοινωνικό πρόβλημα δημιουργεί ένα μεγάλο κόστος σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την κοινωνία μας και υπήρξαν πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για να ποσοτικοποιηθεί το κόστος αυτού του φαινομένου. Μελέτες σε χώρες όπως η Φιλανδία, η Ιρλανδία και κάτω χώρες θεωρούν ότι το κόστος για κάθε άτομο το οποίο αποχωρεί προώρος οδηγεί σε ένα κόστος ενός με 2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο σαν συνολικό κόστος κοινωνικών παροχών κτλ. Αυτό σημαίνει έχουμε ένα, ένα ποσό της τάξης των 30.000 ευρώ το χρόνο για κάθε τέτοιο άτομο και πολλοί θεωρούν ότι αυτό <clears throat> υποτιμά την πραγματικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι αν έχουμε υψηλό επίπεδο πρόλης αποχώρησης σε όλη την Ευρώπη, αυτό θα εμποδίζει την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων όπως είναι η απασχόληση και η διαβίω εκπαίδευση, η κοινωνική συνοχή η στρατηγική για την ευφυά και περιεκτική ανάπτυξη της Ευρώπης 2020. Όχι μόνο λόγω του αντικτύπου που ανέφερα προηγουμένως, αλλά επίσης και οι προβλέψεις για την αγορά εργασίας στην Ευρώπη θεωρούν ότι στο μέλλον μία μόνο για από κάθε δέκα θέσεις εργασίας θα είναι προσβάσιμη στα άτομα αυτά που έχουν φύγει νωρίς από το σχολείο η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό υπήρξε στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την δεκαετία του 1990, αλλά η πιο έντονη εστίαση ξεκίνησε το 2001 όταν θεσπίστηκε κάποιο στόχος και έκτοτε υπήρξαν διάφορες ανακοινώσεις <clears throat> και κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση των νέων που έχουν τονίσει τη σημασία του προβλήματος και πρόσφατα η Κομισιόν παρουσίασε μια πρόταση για ένα σχέδιο δράσης για το ζήτημα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει και τα κράτη-μέλη, ιδίω μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Προγράμματος για τη Διαβίου Μάθηση. Και υπήρξαν και δραστηριότητες μάθησης μεσομοτήμων και ευρωπαϊκά εργαλεία όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δημιουργίας Προσόντων που συνέβαλαν σε αυτή τη διαδικασία. Ποια είναι η κλίμακα τώρα του προβλήματος. Προς το παρόν ένας από κάθε, ένας τους 7 Ευρωπαίους μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αποχωρήσει πρόωρα από το σχολείο. Παλιότερα ήταν περίπου ένας στους 6. Το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ οξύ σε πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης, αλλά επίσης και στο εσωτερικό των μεγάλων αστικών συμπλεγμάτων στη Δυτική Ευρώπη. Πολλές χώρες που βρίσκονται σε καλή θέση είναι μερικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπως η Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία και Σλοβενία. Γενικά, όπως είπα, υπάρχει μία μείωση στο ποσοστό πρόορης αποχώρησης, αλλά η πρόοδος δεν είναι τόσο ταχεία όσο θα θέλαμε. Και στις ε, χώρες της Βόρειας Ευρώπης έχει αυξηθεί αυτό το ποσοστό πρόσφατα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν χώρες όπως το Λουξεμβούργο ή η Λιθουανία όπου μειώθηκε άρδιν αυτό το ποσοστό πρόορης αποχώρησης. Ποιοι τελικά πλήττονται από αυτό το πρόβλημα και γιατί <clears throat> θα πρέπει να τονίσουμε καταρχήν ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολύπλοκο και το οποίο είναι αποτέλεσμα μιας διαργασίας Δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει μετά από μια συγκεκριμένη απόφαση ένα γεγονός. Υπάρχει μια πλειάδα παραγόντων που επηρεάζει την απόφαση για την αποχώρηση και μερικοί από αυτούς τους παράγοντες συνδέονται με τα εκπαιδευτικά συστήματα και μερικά, μερικοί παράγοντες έχουν να κάνουν με εξωγενείς παράγοντες, έχουν να κάνουν με προσωπικές συνθήκες, οι οικογενειακές συνθήκες, οικονομικό πλαίσιο, και <clears throat> περίγυρο των ατόμων που αποχωρούν από το σχολείο. Δεν υπάρχει ένα τυπικό άτομο το οποίο φεύγει πιο νωρίς από το σχολείο, αλλά είναι πιο πιθανό να γίνει αυτό για τα αγόρια, για, τα, για τους μαθητές από μετακινούμενες κοινότητες, από αυτούς που έχουν δύσκολη, ένα δύσκολο οικογενειακό πλαίσιο κτλ. Τι κάνουν τώρα τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Μπορούμε να παρουσιάσουμε τρία είδη απαντήσεων. Στρατηγικού χαρακτήρα προσεγγίσεις, προληπτικές και θεραπευτικού χαρακτήρα για να επανενσωματωθούν αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει νωρίς από το σχολείο. Σε επίπεδο στρατηγική, συντονισμό πολιτικών, καλύτερη συλλογή στοιχείων για να βελτιωθεί η χάραξη πολιτικής σε επίπεδο πρόληψης υπάρχουν είτε στοχευμένες ενέργειες για τους νέους οι οποίοι είναι ομάδα κινδύνου για τα θέματα αυτά και οι απαντήσεις οι οποίες έχουν σε στόχο να βελτιώσουν γενικά το εκπαιδευτικό σύστημα και επομένω να μειώσουν τον κίνδυνο πρόορης αποχώρησης. Και επίσης η επανεσωμάτωση γίνεται με μέτρα τα οποία έχουν σαν στόχο να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία για αυτούς που ήδη έχουν φύγει από το σχολείο. Έχουν γίνει πολλές αναλύσεις αυτών των ε, μέτρων και έχουμε πολλά παραδείγματα τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεσή μας, περίπου 180 διαφορετικά παραδείγματα από τα 27 κράτη-μέλη. <clears throat> Μπορεί να σας ενδιαφέρει λοιπόν να το διαβάσετε αυτό. Σε γενικές γραμμές αν δούμε ποια είναι τα θετικά στοιχεία της προσέγγισης των κρατών μελών για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Μεταξύ αυτών με τους οποίους κάναμε συνεντεύξεις υπάρχει εντύπωση ότι σε πολλές χώρες υπάρχει μια στεναρή πολιτική θέληση να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. 43% των ατόμων με τα οποία είχαμε συνεντεύξεις θεωρήσαν ότι υπήρχε πραγματικά μια έντονη πολιτική δέσμευση. Μόνο 20% την χαρακτήρισαν ασθενική αυτή τη δέσμευση. Αλλά πολλές φορές η δέσμευση αυτή θεωρήθηκε ότι δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη και την αναγκαία χρηματοδότηση. Επίσης, θεωρούμε ότι υπάρχει μια μετατόπιση στον τρόπο που αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό από τα διάφορα κράτη-μέλη. Για πολλές χώρες υπάρχει πολύ περισσότερο συντονισμός για τι αρχέ και του τομεί πολιτική που εμπλέκονται στη ζωή των νέων και σε πολλές χώρες υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία σε ένα σαφές πλαίσιο για την αντιμετώπιση της προώρησης αποχώρησης που αποδίδει καρπούς. Βλέπουμε επίσης ότι είναι πολύ θετικό το ότι υπάρχει μεγαλύτερη αναγνώριση της σημασίας του φαινομένου της αποχώρησης. Πολλές χώρες προσπαθούν να παρέμβουν εγκαίρως για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό, να αποτρέψουν λοιπόν την πρόορη αποχώρηση προτού καν εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα. Σε πολλές χώρες σημαίνει ότι υπάρχει καλύτερη προσχολική παιδεία για τα παιδιά και επομένως τα παιδιά ξεκινούν την ε, σχολική εκπαίδευση σε επίπεδο μεγαλύτερης ισότητας. Επίσης για την επανενσωμάτωση αυτών που έχουν αποχωρήσει από το σχολείο <clears throat> υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι γίνεται πιο δύσκολη και πιο πολυδάπανη αυτή η διαδικασία. Όσο πιο νωρίς έχει φύγει το άτομο από το σχολικό σύστημα, επομένως θα πρέπει η αντιμετώπιση να γίνει το ταχύτερο δυνατόν και έχουμε πολλά παραδείγματα χωρών οι οποίες έχουν εισαγάγει επιτυχείς πολιτικές στον τομέα αυτό. Μία άλλη πτυχή τώρα και μιλάμε πάλι για τα δυνατά σημεία αυτής της προσέγγισης. Πολλές χώρες έχουν δοκιμάσει διάφορες ε, επιλογές και έχουν βρει επιτυχείς φόρμουλες για την αντιμετώπιση της επανενσωμάτωσης μέσω ε, λύσεων που έχουν βασίζονται σε μικρές ομάδες με αλληλοϊποστήριξη, με καλύτερη δυνατότητα παροχής συμβουλών και με τη δημιουργία μιας θετικής ατμόσφαιρας, ενός θετικού κλίματος που προωθεί την εμπιστοσύνη μεταξύ μαθητών και καθηγητών. <clears throat> Υπάρχουν επιπλέον στοιχεία που δείχνουν πότε υπάρχει μεγάλη επιτυχία. Βέβαια υπάρχει μια πρόκληση για όλες τις χώρες που ακολουθούν τέτοια προγράμματα να, προγράμματα να έχουν αρκετές θέσεις και αρκετή χρηματοδότηση γιατί πολλές φορές υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση παραπαροχή ευκαιριών. Υπήρξαν μερικά άριστα παραδείγματα τα οποία δίνουν θετικά αποτελέσματα για χώρες και περιοχές, προγράμματα παροχής συμβουλών που ήταν πολύ θετικά σε χώρες όπως οι κάτω χώρες παραγωγής χάρη υπήρξε <clears throat> θετικό αποτέλεσμα από τα κίνητρα, από τα χρηματικά κίνητρα που δίνονται στα σχολεία για να μειωθεί η πρόοδη αποχώρηση και επίσης καλύτερη παροχή συμβουλών και υποστήριξη σε σχολεία επαγγελματική κατάρτισης που μειώνει το ποσοστό αποχώρησης. Κάτι ακόμα το οποίο είναι σημαντικό για αυτούς οι οποίοι εργάζονται στον εκπαιδευτικό τομέα και το έχουν τονίσει κατά σειρώη, αναφερόμενοι στα προβλήματα της ε, σχολικής εκπαίδευσης, έχουν τονίσει πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη, η ενθάρρυνση, η δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος στο σχολείο και στα συστήματα επανενσωμάτωσης για αυτούς οι οποίοι κινδυνεύουν να φύγουν από το σχολείο ή για αυτούς που έχουν ήδη αποχωρήσει. Θέλουν να τονίσουν λοιπόν τη σημασία του να υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για όλους τους μαθητές από όλα τα στρώματα του πληθυσμού. Και η έννοια ότι πράγματι ανήκουν σε ένα σύνολο αυτοί οι μαθητές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια έρευνα περίπου χιλίων μαθητών στη Φιλανδία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση του σχολικού περιβάλλοντος και η ενθάρρυνση της αίσθηση ότι ανήκει κανείς στο περιβάλλον του σχολείου ήταν ο πιο αποφασιστικός παράγων. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε θετική απόκριση παρά το γεγονός ότι <clears throat> υπήρξε διαφορετική άποψη μεταξύ των κρατών μελών, θεωρήσαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο, γιατί τους έδωσε δυνατότητα να ξεκινήσουν δράσεις και να προωθήσουν δράσεις για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Περίπου το 2 τρίτα αυτών με τους οποίους κάναμε συνεντεύξεις θεώρησαν ότι ο στόχος του 10% έχει οδηγήσει σε θετικές πολιτικές στη χώρα τους. Τους βοήθησε, γιατί έχει βοηθήσει να είναι πιο ορατό αυτό το πρόβλημα. Πού βρίσκονται τώρα οι αδυναμίες για τα θέματα αυτά. Καταρχήν υπάρχει ακόμα κατακαιρματισμός και ανεπαρκής συντονισμός για τα θέματα αυτά. Το 1 τρίτο των εμπειρογνωμών μας θεώρησε ότι δεν υπήρχε αρκετό συντονισμός, ότι ήταν ασθενικός ή προβληματικός ο συντονισμός. Επίσης, <clears throat> πολλές φορές η εστίαση είναι σε συγκεκριμένα σχέδια μονάχα και όχι στην αλλαγή της νοοτροπίας και του τρόπου εργασίας των αρχών και επίσης ε, το σχολικό πρόγραμμα στο, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν θεωρήθηκε ότι δίνει αρκετές ευκαιρίες για πολλούς νέους και ότι δεν δίνει αρκετή εστίαση στις απαραίτητες δεξιότητες. Περαιτέρω <clears throat> αρνητικά σημεία ήταν ότι δεν υπήρχε προσωπικοποιημένη υποστήριξη, δεν υπήρχε αρκετή, δεν υπήρχε αρκετή διαβούλευση με τους νέους κτλ. Ποιες είναι τώρα οι συστάσεις μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της πρόορης αποχώρησης ως ένα πολύπλοκο θέμα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μονάχα από τους εκπαιδευτικούς ή από τις εκπαιδευτικές αρχές. Υποστηρίζουμε επίσης τη συνέχιση της παρακολούθησης των εξελίξεων σε σχέση με την διάσταση και το εύρος αυτού του φαινομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να παροτρύνουμε και τα κράτη-μέλη να το πράξουν επίσης. Είναι πολύ θετικό επίσης το να υπάρχει ανταλλαγή ε, πρακτικών και πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και με καλύτερη εστίαση και στόχευση μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Η συγκρηματοδότηση είναι κάτι το οποίο το έχουν ζητήσει τα κράτη-μέλη του τον τομέα αυτό και η πρότασή μας για τα θέματα αυτά θα ήταν να δοθεί περισσότερη προσοχή στο μέλλον για τα κριτήρια επιλογής ώστε να υπάρχει μια πολυκλαδική προσέγγιση και να τροποποιηθούν οι κρατούσες πρακτικές και όχι μονάχα να προχωρούμε σε νέα σχέδια για τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές. <clears throat> Οι συστάσεις μας είναι ότι οι χώρες που έχουν ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και βασίζονται σε στοιχεία αριθμητικά από τη βάση των οποίων χαράζουν πολιτική. Αυτό είναι πολύ θετικό. Επίσης πρέπει να υπάρχει μια περιεκτική προσέγγιση για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής που λαμβάνει υπόψη αυτούς οι οποίοι είναι εμπλεκόμενοι αλλά και τις απόψεις των μαθητών, τα ερευνητικά στοιχεία και την αλληλεπίδραση με άλλες πολιτικές. Θα ήταν χρήσιμο πέρα της συνεργασίας να υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει την κεντρική ευθύνη για την εφαρμογή αυτών των σχεδίων. πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί και η σωστή ισορροπία <clears throat> μεταξύ της ε, πρόληψης της, ε, και της, ε, του μετριασμού της μείωσης του προβλήματος αυτού και της επανεσωμάτωσης και κυρίως να υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για όσους θέλουν να επανερθούν στο σχολείο. <clears throat> Μέσα στην περιεκτική τώρα αντιμετώπιση για την ανάπτυξη των πολιτικών, θεωρούμε επίσης ότι είναι απαραίτητο να, να βασιστούμε και στην εμπειρία των νέων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινωνικών εταίρων κτλ. Επίση, οι γονεί θα πρέπει να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και είναι χρήσιμο τα σχολεία να δίδουν περισσότερα εργαλεία <clears throat> μαζί με τους ε, με μεγαλύτερη συνεργασία με τους γονείς των παιδιών που κινδυνεύουν να αποχωρήσουν από το σχολείο. Χρήσιμο είναι επίσης να υπάρχουν τοπικές λύσεις στα τοπικά προβλήματα και αυτό είναι πολύ θετικό. Εν κατακλείδη ορισμένα στοιχεία τα οποία ανέφερα και προηγουμένως, να υπάρξει και κάποια αναθεώρηση σε ορισμένα πλαίσια του σχολικού προγράμματος στο δεύτερο βάθμιο επίπεδο, να βοηθηθούν με πρόσθετα μαθήματα οι μαθητές οι οποίοι <clears throat> υπολείπονται των υπολείπων. Παραδείγματος χάρη μία έρευνα στην Ισπανία περίπου 900 ατόμων που αποχώρησαν από το σχολείο έδειχνε ότι ο ένας από τους 9 έφυγαν γιατί χρειάστηκε, ε, έμεινα μεταξυταστέ και πρέπει να ξανακάνουν έπρεπε να επαναλάβουν μάλλον ένα χρόνο και αυτό ήταν μια πολύ κακή εμπειρία για αυτούς. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο και για την παροχή συμβουλών, ιδίως στα σημεία καμπής από <clears throat> την αρχή της δευτεροβάθμιας ε, εκπαίδευσης στο δεύτερο τμήμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι πολλές φορές ένα σημείο στο οποίο υπάρχουν απώλειες μαθητών. Σας ανέφερα επίσης τη σημασία του να έχουμε ένα θετικό περιβάλλον στο σχολείο και μεγάλες προσδοκίες για όλους. Κάτι ακόμα το οποίο είναι σημαντικό είναι και η υποστήριξη των διδασκόντων. Δεν είναι πιο εύκολο το έργο των διδασκόντων και υπάρχουν πολλές ε, αιτήσει να υπάρξει μεγαλύτερη υποστήριξη από τους διδάσκοντες για τους μαθητές οι οποίοι κινδυνεύουν να αποχωρήσουν. Αυτό σημαίνει όμως περισσότερη υποστήριξη και εκπαίδευση των διδασκόντων για να μπορέσουν να έχουν και αυτό τον ρόλο. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω για την έρευνα αυτή. Έχουμε πάρα πολλά πορίσματα. 300 σελίδες περίπου είναι η έκθεσή μα Και έχουμε και μια άλλη έκθεση η οποία είναι υπό προετοιμασία. Θα την ε, διανύμουμε στις επόμενες μέρες και αν υπάρχουν ερωτήματα με μεγάλη χαρά θα προσπαθήσω να απαντήσω. Είμαι η μόνη που είμαι εδώ από την ε, ομάδα μας αν δεν μπορώ να απαντήσω τα ερωτήματά σας, όμως θα επανέλθω γραπτός αφού συζητήσω με τους συναδέλφους μου. Thank Η πρόεδρος ΠΑΚ, σας ευχαριστώ πολύ, ανάψτε τα φώτα. Ευχαριστώ. Κυρία Νεβάλα, πολύ περιεκτική η παρουσίαση δείχνει πόση πολλή δουλειά κρύβεται από πίσω. Ευχαριστώ και τα πρόσωπα που έψαξαν και σας βρήκαν, γιατί δεν είναι και πάντα εύκολο να βρεθούν τα σωστά πρόσωπα και ασφαλώς η μελέτη σας θα βοηθήσει πολύ στην εργασία μας. Αν έχουμε το στόχο να κατέβουμε μέχρι το 2020 από τα 15% στα 10% θα χρειαστεί βέβαια πολύ μεγάλη προσπάθεια και εσείς μας προσφέρατε πολλές ιδέες, μας δώσατε υποδείξεις για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Η κυρία Χάνιμπαλ είναι η συγγήτρια για το θέμα και ασφαλώς θα προσφύγει στα πορίσματά σας, στην ε, έκθεσή σας, στην εργασία της, δηλαδή στην έκθεσή της. Εμείς αναθέσαμε τη μελέτη αυτή ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα πολύ όμως να λάβει υπόψη την έκθεση αυτή, μάλλον τη μελέτη σας αυτή, ε, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί νομίζω ότι θα διευκολύνει το έργο, το έργο των αρμοδίων. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνει επικάλυψη έργου αφού ήδη έχει γίνει μία φορά η μελέτη. Θα αρχίσουμε τώρα την συζήτηση και θα παρακαλέσω τις συναδέλφους και τους συναδέλφους είτε να κάνουν ερωτήσεις είτε να κάνουν σχόλια. Ο κύριος Καβαντά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εσάς και την ομάδα σας για αυτήν την έκθεση που αποτελεί και τη βάση των σχέσεων που θα θέλαμε να διατηρήσουμε με την ομάδα σας γιατί έχετε συντάξει την πρώτη μελέτη που υπάρχει σχετικά στην Ευρώπη. Μιλήσατε για το κόστος της εγκατάλειψης του σχολείου, ένα εκατομμύριο ευρώ. Τι σημαίνει, είναι ένα κοινωνικό διαβίου κόστος ή είναι το κόστος μη εξελίξιμης σταδιοδρομίας, είναι το κόστος της κατάρτισης, το κόστος της κοινωνικής προστασίας. Τι αντιπροσωπεύει αυτό το κόστος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Ευχαριστώ που, που συντάξατε αυτήν τη μελέτη για ένα θέμα τόσο σημαντικό. Πάμε τώρα στο θέμα που με ενδιαφέρει στην παρουσίασή σας επιμείνατε στο γεγονός ότι θα πρέπει να εξατομικεύσουμε τον τρόπο διδασκαλίας, να δημιουργήσουμε θετική ατμόσφαιρα κλπ. Τώρα ξέρετε όμως ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω λιτότητας ε, έχουμε την τάση να δημιουργούμε σχολικές τάξεις με ολοένα παραπάνω μαθητές. Με άλλα λόγια, όλα όσα αφορούν στις υποχρεώσεις μας διδασκαλίας και ε, παιδείας ε, περιορίζονται σε αυτή τη φάση των ισχνών αγελάδων. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Τι σκέφτεστε εσείς για αυτή την εξέλιξη. Και να επανέλθω τώρα στους δασκάλους. Πρέπει να, να είναι ειδικευμένοι. Ο ρόλος τους είναι βασικότατος, είναι θεμελιώδης. Κατά τη γνώμη σας, λαμβάνουμε επαρκώς υπόψη την σημασία της κατάρτισης των διδασκόντων στην Ευρώπη. Έχουμε επαρκείς εξειδικευμένους δασκάλους. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βέρ. Και εγώ ευχαριστώ την φιλοξενούμενη μας για αυτήν τη μελέτη. Σήμερα συζητάμε μία έκθεση πάρα πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την συνεισφορά μίας εμπειρογνωμονός. Και θέλω να ευχαριστήσω και την Κομισιόν για το στόχο που όρισε της μείωσης δηλαδή της εγκατάλειψης του σχολείου στο 10%. Φαντάζομαι ότι μπορούμε όμως να εξυγχρονίσουμε και τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη. Εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία βρίσκονται υποπίεση στην Ευρώπη δεν υπάρχουν πια νέοι. Είμαστε μια γερασμένη κοινωνία, αλλά από την άλλη μεριά το 1 πέμπτο των νέων μας δεν έχουν δουλειά και πολλοί νέοι βρίσκονται εκτός σχολικού συστήματος. Αυτό είναι μια καταστροφή. Οι νέοι που είναι λίγοι στην Ευρώπη δεν καταφέρνουν να ενσωματωθούν σωστά στην κοινωνία. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την πίεση, να εξυγχρονίσουν τα σχολεία και ή δυνατόν να δώσουν μια δεύτερη ή και τρίτη ευκαιρία στους νέους. Δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε ούτε ένα νέο και να τον, στην Ευρώπη και να τον αφήσουμε εκτός σχολικού συστήματος. Είδαμε εμείς ε, ποιο είναι το κόστος ε, των, ε, που υπολογίζουν οι οικονομολόγοι. Πρόκειται για ένα τεράστιο οικονομικό κόστος. και από τη δική μου πλευρά σας ευχαριστώ για τη μελέτη σας. Είχα κάνει γνωμοδότηση για την Επιτροπή Απασχόλησης και χαίρομαι που τώρα μπορούμε να φωτίσουμε το θέμα από άλλη σκοπιά. Και βέβαια στην Επιτροπή Απασχολήσεως είχαμε διαπιστώσει ότι ένα μεγάλο δυναμικό μένει άπραγο. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι η προληπτική ας πούμε προσέγγιση να αποφευθεί δηλαδή η εγκατάλειψη του σχολείου και επ' αυτού σίγουρα όπως είπε ο κύριος Τάκουλα θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε την ε, μάθηση, τη διδασκαλία πιο εύκαμπτη και πιο προσαρμόσιμη στις ε, ατομικές ανάγκες. Έχετε στη μελέτη σας εξετάσει την προληπτική προσέγγιση. Γιατί σε πολλές χώρες υπάρχει μια πολύ περιοριστική και μάλλον κατασταλτική νοοτροπία, δηλαδή στέλνουν την αστυνομία να πάει τα παιδιά με το ζόρι στο σχολείο. Όταν όμως δεν πηγαίνει ο τη κάθε μέρα στο σπίτι του παιδιού να το πάρει να το πάει στο σχολείο, πάλι σταματάει το παιδί να πηγαίνει στο σχολείο. Έχουμε λοιπόν ε, τέτοια ε, παραδείγματα. Έχετε κάνει κάποια μελέτη και έχετε ποσοστά. Η κυρία Βενεραπάτου. Ευχαριστώ. Εγώ ενδιαφέρθηκα για τα, στη θέση των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο. Και γιατί εγκαταλείπουν τα παιδιά το σχολείο, γιατί έχουν κακά αποτελέσματα. Λένε εντάξει έχω κακούς βαθμούς, φεύγω υποχρεώνουμε τους μαθητές, ε, να είναι, ε, αξιολογούμε μάλλον τους μαθητές στην, πώς κάθονται στην τάξη, πολλές ώρες ε, ακίνητοι ή αξιολογούμε τελικά τις γνώσεις και τις ικανότητες. Διότι αν βαθμολογούμε τις γνώσεις και τις ικανότητες πρέπει να δούμε και ποια είναι η παιδαγωγική προσέγγιση. Θα πρέπει να σκεφτούμε ποιος είναι ο τρόπος διδασκαλίας και εκμάθησης. Βλέπουμε ότι πολλά παιδιά είναι πιο πολύ ε, ακουστικοί τύποι ή οπτικοί τύποι και αφομοιώνουν καλύτερα κατά αυτόν τον τρόπο. Και θα έπρεπε Για να μπορέσει κάποιος πραγματικά να έχει κέφι να μάθει ε, πρέπει να του δίνεται και η δυνατότητα. Εγώ είμαι κόρη, εργάτη, γεννήθη, έρχομαι από την Αλγερία, ε, έζησα στα λαϊκά στρώματα. Νομίζω ότι το παιδαγωγικό σύστημα είναι ουσιαστικό για να κρατήσει τους νέους. Είχα την ευκαιρία να πάω στη Γερμανία και είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Πρέπει κανείς να είναι ιδιαίτερα δυναμικός στη φάση της εκμάθησης. Πολλές φορές ε, τα παιδιά τα οποία εγκαταλείπουν το σχολείο λαμβάνονται, λαμβάνονται υπό, την υπό την κοινοτική προστασία μέσα από η ίδια η κοινότητα τους βοηθάει στη διαδικασία της εκμάθησης. Εγώ αυτό το οποίο έζησα στη Γαλλία στα σχολικά μου χρόνια αλλά και μετά όταν συνέχισα να παρακολουθώ τα πράγματα διαπίστωσα ότι το σημαντικό ήταν το να μαθαίνει κανείς την μάθηση να μαθαίνει πώς μαθαίνει. Και τι άλλο ήθελα αλήθεια να πω. Τώρα νομίζω επίσης ότι για να έχει κανείς και το σχετικό πνεύμα έναντι της γνώσης πρέπει να είναι και απολευθερωμένος από κοινωνικές, ψυχολογικές πιέσεις, αν ένα παιδί έχει ψυχολογικά προβλήματα, έχει αισθηματικά προβλήματα, έχει κοινωνικά προβλήματα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη γνωστική διαδικασία. Χρειάζονται λοιπόν πολλαπλές ομάδες εκμάθησης, παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, γιατροί, να έχουμε μία ομάδα ολοκληρωμένη που να επιτρέπει μία ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος και να εγγυάται και την προσωποποιημένη παρακολούθηση. Θα πρέπει επίσης να έχουμε και μία ε, συνοδεία του μαθητή για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Πρέπει να έχει μία προβολή στο μέλλον ο νέος, γιατί άμα δεν την έχει τότε εγκαταλείπει τον εαυτό του. Και επίσης και το διδακτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο. Η ε, Πακ, πρόεδρος. Ευχαριστώ. Έχω και μία παρατήρηση. Α, αυτός ο στόχος που έχουμε, δηλαδή μείωση των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο, χρειάζεται και διαφορετική κατάρτιση των δασκάλων. Αυτό μου φάνηκε να λείπει λίγο στη μελέτη σας. Το ζήτημα δεν είναι να μεταφέρουν μονάχα την γνώση των βιβλίων. Να πάρουν το παιδί εντό εισαγωγικών από το χέρι, από εκεί που ξεκινά και να το καθοδηγήσουν σε όλο το δρόμο μέχρι να γίνει πλέον αυτόνομο. Το γεγονό ότι έχουμε και όλο λιγότερα παιδιά, ίσω αυτό να έχει ένα πλεονέκτημα με την έννοια ότι έχουμε περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούμε με το μεμονωμένο παιδί, να προαγάγουμε τη δημιουργικότητά του, τα παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο δεν σημαίνει ότι δεν έχουν καμία ικανότητα ή δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν εάν τα βοηθούσαν κάποιοι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πρώτον δασκάλους που να μπορούν να το κάνουν αυτό, επίσης περισσότερους κοινωνιολόγους, παιδαγωγούς που θα μπορέσουν να εγκύψουν περισσότερα στα προβλήματα των παιδιών, ώστε να έχουμε για καλύτερα καταρτισμένους ανθρώπους εν τέλει για την αγορά εργασίας. Και χρειαζόμαστε και ένα ουσιώδες περιεχόμενο που να είναι περισσότερο κομμένο και αραμένο στις ανάγκες του καθενός. Στην τελευταία συνεδρίασή μας εδώ, ο πρόεδρος Λόθαρ Μπίσκι είχε πει ότι πρέπει να προσέξουμε τα παιδιά να οδηγούνται σε επαγγέλματα τα οποία να είναι σημαντικά, αλλά που δεν είναι απαραίτητο να έχουν την ε, ε, σούπερ ειδικότητα. Για παράδειγμα, ο υποδηματοποιός Τη γειτονιά, Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που στην ε, περιοχή μου έχω έναν καλό τσαγκάρι ο οποίο διορθώνει σωστά τα παπούτσια. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά βέβαια μπορούμε να τα λέμε αυτά, μπορούμε εδώ να τα λέμε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Γι' αυτό χαίρομαι, ή τουλάχιστον δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε μόνοι μα, γι' αυτό χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ευθυγήσει τις ιδέες αυτές και ίσω μπορεί να βοηθήσει ώστε να προωθήσουμε τις βέλτιστες αυτές πρακτικές. Αυτά από την πλευρά μου. Θα δώσω το λόγο πάλι στην κυρία Νεβάλα να, να απαντήσει και μετά θα λάβει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Αν Μαρή Νεβάλα. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια καθώς και για τις ερωτήσεις σας. Συμφωνώ απολύτως με τα θέματα που θέσατε και νομίζω ότι τα θίγει η έκθεσή μας. Η πρώτη ερώτηση τώρα για το κόστος. Οι μελέτες τις οποίες αναφέρθηκα και που είναι τρεις ξεχωριστές μελέτες από ξεχωριστές χώρες είναι λοιπόν λίγο διαφορετικές κατά τη μεθοδολογία τους αλλά βέβαια πάντα περιλαμβάνουν το κόστος που είναι ε, υπολογισμένο στη βάση του απολεσθέντος εισοδήματος. Από την εκπαίδευση αυτή θα επέστρεφε 70.000 ευρώ ο κάθε μαθητής στη διάρκεια της ζωής του. Χάνονται και έσοδα φορολογικά. Ορισμένες από τις μελέτες αυτές περιλαμβάνουν και το στοιχείο που συνδέεται με την εγκληματικότητα καθώς και με την υγεία, διότι πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι παιδιά που εγκαταλείπουν νωρί το σχολείο δυστυχώς πολύ συχνά πέφτουν σε εγκληματικές ενέργειες. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο τώρα για το μέγεθος των σχολικών τάξεων, των αιθουσών δηλαδή και των δασκάλων. Αυτό μας ανησύχησε πολύ, αλλά ανησυχεί πολύ και πολλούς από τους ανθρώπους με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή. Πήγαμε σε χώρες όπου έχουν αυξήσει τη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση της ε, προήμιση κατάληψη του σχολείου. Αλλά από την άλλη μεριά έχουν μειώσει τις δαπάνες για ειδικέ εκπαιδεύσεις. Και αυτό είναι πρόβλημα, διότι ορισμένοι θεωρούν ότι αν περικόπτονται αυτές οι βασικές υπηρεσίες, θα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για ειδικέ ε, πολιτικές μετά για το θέμα αυτό. Το μέγεθος των τάξεων είναι βέβαια μέγα θέμα και πολύ σημαντικό με, κυρίως με νεαρά άτομα τα οποία ε, βρίσκονται σε κίνδυνο να περάσουν σε εγκληματικές ε, ενέργειες και συχνά διατίθεται χρηματοδότηση για σχολεία σε ορισμένες περιοχές για να μειωθεί το μέγεθος των τάξεων Συνήθως απαιτείται πάντως μια δέσμη μέτρων η οποία θα συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων. Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των δασκάλων, δεν το εξετάσαμε βέβαια με λεπτομέρεια, αλλά όταν μιλήσαμε με τα αρμόδια πρόσωπα, βρήκαμε πολύ λίγα παραδείγματα που να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα αυτό είτε με διαρχή κατάρτιση είτε με άλλο τρόπο. Για την ώρα δεν έχουμε στοιχεία που να δείχνουν ότι θα υπήρχε αύξηση για την κατάρτιση των δασκάλων για τέτοια θέματα. Και αυτό το έθεσαν βέβαια ως θέμα και οι εκπρόσωποι των δασκάλων με τους οποίους μιλήσαμε για το θέμα τώρα, εάν μπορεί κανείς να εξαναγκάσει τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Στις χώρες που εξετάσαμε δεν, είχαμε, δεν είδαμε παραδείγματα χρήσης των αστυνομικών δυνάμεων για να πάνε τα παιδιά με το ζόρι στο σχολείο. Άκουσα βέβαια ότι υπάρχουν τέτοιες πολιτικές, δεν θυμούμαι αν ήταν στην Γερμανία ή ίσως εδώ στο Βέλγιο, αλλά δεν το γνωρίζω, δεν γνωρίζω δηλαδή εγώ προσωπικά εγώ προσωπικά και η ερευνητική μου ομάδα και τα στοιχεία που συλλέξαμε δείχνουν ότι δεν μπορεί κανείς να αναγκάσει κάποιον να μάθει. Πρέπει να εξευρεθούν οι σωστές εναλλακτικές επιλογές για το συγκεκριμένο νεαρό πρόσωπο. Ορισμένοι που έχουν δουλέψει, κάτι μάλλον που έχει αποδώσει σε ορισμένες χώρες είναι να δοθεί μια ευκαιρία να δοκιμάσει το παιδί διάφορες επαγγελματικές ε, καταρτήσεις για διάρκεια ενός έτους. Να ψάξουμε δηλαδή να βρούμε τι ακριβώς ενδιαφέρει το συγκεκριμένο παιδί, τι του αρέσει. Τέτοιου είδους πολιτικές αποδείχθηκαν χρήσιμες γιατί προσφέρουν στους νέους τη δυνατότητα να πάνε για ένα χρόνο και να δοκιμάσουν τελείως διαφορετικά επαγγέλματα μέσω του βρουν κάτι που να τους αρέσει πραγματικά και τότε να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στον τομέα αυτό. Συμφωνώ με τα παραδείγματα που ανέφεραν οι συναδελφοί σας ε, σχετικά με την ανάγκη της καθοδήγησης γιατί αλλιώς οι νέοι, οι νέες θα εγκαταλείψουν το σχολείο. Συμφωνώ επίσης και με τη σημασία του counseling, δηλαδή της παροχής συμβουλών, καθώς και για την καλύτερη εκατάρτιση των δασκάλων. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Άνταμ Πορκόνη. Μερσή κύριε Πρόεδρε, δύο-τρία σχόλια. Τα ουσιαστικά θα τα δείξω στη συνέχεια που θα γίνει η συζήτηση επί του θέματος ημερησίας διάταξης. <clears throat> Τονίστηκε ότι το θέμα αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες για τη σύνολη Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το στόχο του 10% για το επίπεδο του 2020 τον προηγούμενο Ιούνιο και υπάρχει το πακέτο αυτό για την ανακοίνωση αυτή που αφορά την αντιμετώπιση της πρόορης απασχόλησης από το σχολείο. Υπάρχει και ένα έγγραφο εργασίας που περιέχει πολλά παραδείγματα και ανάλυση και υπάρχει και η πρόταση για μια σύσταση του Συμβουλίου. Η σύσταση αυτή τώρα έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο. Το σύνολο πακέτου, το σύνολο πακέτο μάλλον υποστηρίχθηκε ιδιαίτερα από το Συμβούλιο. Και η σύσταση κρίθη τον προηγούμενο μήνα στο Συμβούλιο Παιδείας. Τα κράτη-μέλη όμως που είναι τα αρμόδια για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό, που έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα, προσβλέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τους βοηθήσει να διδαχτούν από τις βέλτιστες πρακτικές, να γνωρίσουν τι συμβαίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρχει κατάλληλη γνώση και έρευνα για τα θέματα αυτά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε λοιπόν το Κοινοβούλιο που ζήτησε να συνταχθεί αυτή η έκθεση. Ευχαριστούμε και την Αν Μαρή και την ομάδα της που μας δίνουν κάτι που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την ε, ανάλυση αυτή. Θα δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασία σε επίπεδο κρατών μελών για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή και ιδίως να παρακολουθήσουν τις δεσμεύσεις των κρατών μελών για να υπάρχουν πλήρεις εθνικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσετε η πρώην σχολική αποχώρηση. Θα το κάνουμε αυτό μέχρι το 2012 και η τελική έκθεση με την ανάλυση αναχώρε και τις συστάσεις θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο Θέλει μια βασική εισρωή σε αυτή τη διαδικασία. Κάτι ακόμα το οποίο θέλω να αναφέρω είναι μια ακόμα έκθεση την οποία έχουμε ε, θέσει στη διαδικασία, έχουμε ζητήσει διαδικασία προσφορα, προσφορών για την εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας, για τις μη παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης για αυτούς οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το σχολείο και να δούμε τι στοιχεία αυτής της ε, έκθεσης μπορούν να συμπεριληφθούν στην στον κύριο κορμό της εκπαίδευσης, γιατί όπως είπαν πολλοί ομιλητές, πρέπει να έχουμε μια πιο στοχευμένη και καλύτερα προσαρμοσμένη προσέγγιση και υπάρχουν ήδη πολύ καλά παραδείγματα για το να δίδεται μια δεύτερη <clears throat> ευκαιρία έξω από τη σχολική εκπαίδευση και πολλοί δεν έχουν χρησιμοποιήσει αυτέ τι ευκαιρίε. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολή προσφορών και θα σα στείλουμε την έκθεση όταν είναι στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ, Αδάμ. <clears throat> Έχουμε κλείσει λοιπόν αυτή τη συζήτηση. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ, αν Μαρία, εσά και του ε, συνεργάτε και συνεργάτηδέ σα. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 8, το οποίο ουσιαστικά αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, αλλά από την οπτική γωνία τη ε, εισηγήτριά μα, τη κυρία Χάνιμπαλ. Έχετε το λόγο, κυρία Χάνιμπαλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ θετική αυτή η ευκαιρία να συντάξω αυτή την έκθεση. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αναλάβει το θέμα αυτό. Είχα ήδη αναλάβει μια έκθεση για την προώρη σχολική προώρη στο παρελθόν και φυσικά υπάρχει ε, μεγάλη επικάλυψη μεταξύ των δύο εκθέσεων. Θέλω να ευχαριστήσω την Αν Μαρή Νεβάλα για την έκθεσή της, η οποία ήταν πάρα πολύ πλήρης και είχα πάρει και πιο νωρί σε ένα προσχέδιο αυτή τη έκθεσης. Πολλά από τα πράγματα που περιλαμβάνει η έκθεσή μου έχουν τροφοδοτηθεί από αυτή τη μελέτη που είναι η ίδια η μόνη μελέτη αυτού του είδου και μα δίνει πάρα πολύ χρήσιμε πληροφορίε. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να δούμε αυτή την παρουσίαση και να μάθουμε περισσότερα για το περιεχόμενο τη έκθεση αυτή. Η πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου είναι μία από τι βασικέ προκλήσει που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2009 πάνω από 6 εκατομμύρια νέοι εγκατέλειψαν τη σχολική εκπαίδευση μόνο με <clears throat> ένα χαμηλό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή λιγότερο. Σχεδόν ένας στους δύο από αυτούς που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο ήταν άνεργος ή εκτός αγοράς εργασίας. Αυτό μας δίνει και μία εικόνα της διάστασης του προβλήματος. Όπως ακούσαμε το 2003 τα κρατη αποφάσισαν να μειώσουν το ποσοστό πρόορης εγκατάλειψης σε λιγότερο από 10% μέχρι το 2010. Δυστυχώς όμως μόνο 7% των κρατών μελών το έχουν επιτύχει αυτό. Υπάρχουν 7 κράτη-μέλη μάλλον το πέτυχαν, αλλά έχουμε άλλα 20 κρατη που πρέπει να το επιτύχουν. Όταν εισήχθη αυτός ο στόχος, αποφασίστηκε ότι η μείωση του ποσοστού πρόορης εγκατάλειψης σε λιγότερο από 10% το 2020 θα είναι ένας από τους κύριους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Είναι πολύ θετικό λοιπόν που η Επιτροπή μας εργάζεται για κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται πολύ θετικά ως ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ως ένας από τους στόχους προς επίτευξη. Μας είπε η έκθεση της κυρίας Νεβάλα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι τρομακτικό όταν αναφερόμαστε στο ένα έβδομο των μαθητών σε σχολικό επίπεδο, όπως συμβαίνει πολλές φορές με αυτά τα θέματα, τα εκπαιδευτικά. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός <clears throat> για την εγκατάληψη. Εγώ χρησιμοποιώ τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάποιος που εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο είναι κάποιος μεταξύ 18 και 24 χρονών που έχει φύγει από το σχολείο με χαμηλό δευτεροβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης ή κάτι λιγότερο. Αυτό είναι και ο ορισμός που χρησιμοποιήθηκε από την ε, κυρία Νεβάλα στην παρουσίαση που σας έδειξε προηγουμένως. Βέβαια δεν υπάρχει ο τυπικός εγκαταλειψίας του σχολείου και δεν υπάρχει και μια στάνταρ προσέγγιση για αυτούς οι οποίοι κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο. Είναι πολύ μορφή αυτή η ομάδα του πληθυσμού και δεν φεύγουν όλοι από το σχολείο για αρνητικού λόγους. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Η χαμηλή ε, απόδοση είναι ένας καλός παράγων για την πρόβλεψη του κίνδυνου πρόορης ε, εγκατάλειψης. Αυτοί λοιπόν που έχουν να αγωνιστούν στη σχολική τους παιδεία πολλές φορές χάνουν το κίνητρο να παραμείνουν στο σχολείο ενώ αυτοί οι οποίοι είχαν ισχυρή ε, ε, εκπαιδευτική απόδοση παραμένουν στο σχολείο παρά όλους τους εξωτερικούς εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη σχολική τους καριέρα. Δεν μπορούμε να δούμε όμως τη χαμηλή απόδοση απομονωμένα γιατί συνδέεται με άλλα στοιχεία όπως είναι η, η ένδια, η κακοποίηση, το, η προέλευση και το ε, κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο μιας οικογένειας και όταν η οικογένεια δίνει ένα σταθερό περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν τα παιδιά να αναπτυχθούν και να μορφωθούν, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα ότι ένα μαθητής θα συνεχίσει τη σχολική του εκπαίδευση. Όταν όμω οι οικογένειε δεν ενθαρρύνουν του νέου <clears throat> να μείνουν στο σχολείο, τότε η προώρια εγκατάλειψη γίνεται πολύ πιο πιθανή. Και υπάρχουν και άλλε ορατέ, άλλοι ορατοί συντελεστέ, Βλέπουμε να υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, ανισότητε σε περιφερειακό επίπεδο και μία διαφορά μεταξύ του χώρου της υπαίθρου και του χώρου των ε, πόλεων. Δεν είναι εκπληκτικό ότι είναι πιο μεγάλο το ποσοστό εγκατάλειψης μεταξύ των μεταναστών πληθυσμών και των εθνοτικών μειονοτήτων, κυρίως μετά τον Ρώμα, μεταξύ των Ρώμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα κύριο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είναι και θέμα φύλου επίσης. Τα κορίτσια <clears throat> είναι πολύ πιο απίθανο να εγκαταλείψουν το σχολείο 13% για τα κορίτσια, 17% για τα αγόρια είναι το ποσοστό πρόορης εγκατάλειψης. Και αυτό λοιπόν πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Εγώ σοκαρίστηκα επίση όταν είδα τα στοιχεία για το τι κοστίζει η σχολική εγκατάληψη. Ένα με δύο εκατομμύρια ευρώ σε μία κατά τη διάρκεια όλη τη ζωή των ατόμων αυτών. Και υπάρχουν φυσικά και άλλε συνέπειε και όχι μόνο οικονομικέ συνέπειε. Όπως ακούσαμε, η πρώτη εγκατάλειψη έχει αρνητική επίπτωση στην κοινωνική ενσωμάτωση και στην οικονομική ευρωστία των ατόμων αυτών. Επομένως μπορεί να ποσοτικοποιήσει κανείς όχι μοναχα κοινωνικά αλλά και οικονομικά το κόστος της πρώτης εγκατάλειψης για τα νέα αυτά άτομα και σε μια εποχή οικονομικών δυσκολιών όχι μονάχα στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο, το οικονομικό επιχείρημα είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό το οποίο θα πρέπει να το υπερτονίσουμε. Θεωρούν πολλοί ότι το να μειωθεί το ποσοστό αυτών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο κατά 1% μονάχα θα δημιουργήσει μισό εκατομμύριο προς, πρόσθετες δυνατότητες απασχόλησης για τους νέους. <clears throat> Και όταν δούμε όσο αυξάνονται οι θέσεις απασχόλησης που απαιτούν υψηλό επίπεδο προσόντων και εκπαίδευσης και πάλι αυτό είναι ένα σημαντικός παράγον. Ξέρουμε ότι και η διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση αυτών που φεύγουν από το σχολείο χωρίς πλήρη προσόντα είναι πολύ πιο περιορισμένη και η έλλειψη εκπαιδευτικών προσόντων πολλές φορές είναι κάτι το οποίο προκαθορίζει την ένδυα στο μέλλον. Αυτοί που τελειώνουν το σχολείο με λιγότερα προσόντα έχουν πολύ λιγότερες επιλογές μέσα στην αγορά εργασίας. Πολλές φορές έχουν επισφαλείς κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας που δεν έχουν μέλλον. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η πρόορη εγκατάλειψη η πρόληψη της πρόληψης εγκατάλειψης μπορούν να σπάσουν τον φαύλο κύκλο της ένδυας από τη μια γενιά στην άλλη και να βελτιώσουν την οικονομική ανάπτυξη. Επίσης έχει και σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, γιατί η πρόορη εγκατάλειψη σημαίνει και υψηλό επίπεδο ε, αντικοινωνικής συμπεριφοράς, πρόορης εγκυμοσύνης και κατάχρησης ναρκωτικών. Όπως ακούσαμε βέβαια δεν είναι απλό το θέμα αυτό, είναι ένα πολύπλοκο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλειών. Δεν υπάρχει μια πανάκια, πρέπει να το δούμε σαν μια δέσμη προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο είναι μια προσωπικοποιημένη αντιμετώπιση, γιατί από ό,τι ακούσαμε υπάρχουν πολλοί παράγοντε που προκαλούν την πρόορη εγκατάλειψη και που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προ το συμφέρον των μαθητών. Αυτό λοιπόν το οποίο προτείνει η εκθεσή μου είναι κάθε σχολείο, κάθε δευτεροβάθμιου επίπεδο σχολείου να έχει και μια υπηρεσία παροχή συμβουλών για να βοηθάει τους μαθητές και οι συμβουλές αυτές να μην είναι μονάχα εκπαιδευτικού χαρακτήρα αλλά να έχουν και ποιμενικό χαρακτήρα σε σχέση με τους μαθητές, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές οι μαθητές έχουν πρόβλημα να πηγαίνουν στο σχολείο και θα πρέπει να ευνοηθούν τα δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν τους μαθητές και δίνουν και συμβουλές και υποστήριξη για την μετέπειτα καριέρα τους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι η χώρα που ξέρω εγώ καλύτερα. Υπάρχει μια οργάνωση που λέγεται η Υπηρεσία Σύνδεσης, η οποία δημιουργήθηκε το 2001, της οποίας ο στόχος να που συνδυάζει την παροχή συμβουλών για το σχολείο και για την καριέρα είναι να δώσει προσωπικοποιημένη υποστήριξη στους νέους έχει εισαγάγει μια σειρά από καινοτομίε. και γενικά θεωρείται ότι έχει κάνει καλή δουλειά <clears throat> και είναι ένας επιτυχής οργανισμός. Κάνει σαφέ επίση η εκθεσή μου ότι η διαδικασία της επανενσωμάτωσης πάλι στον εκπαιδευτικό χώρο θα πρέπει να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατό. Τα προβλήματα ε, από το σχολείο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατό. Γίνονται πιο δύσκολα αν χρονίσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, τόσο το καλύτερο. Πρέπει να δούμε και τις μεθόδους εκπαίδευσης και τις διδακτικές μεθόδους και να ενθαρρύνουμε τα σχολεία να φύγουν από μια μόνο παραδοσιακή διαδικασία δοκιμασιών για τους μαθητές, όπου αυτό είναι απαραίτητο, που κρίνουν τους μαθητές μονάχα σε μια μέρα σε όλο τον χρόνο και να βοηθούν τους μαθητές με μια συνεχή μορφή αξιολόγησης. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί και μεγαλύτερη κινητικότητα μεταξύ διαφόρων σχολικών κατευθύνσεων και να έχουν οι μαθητές τη δυνατότητα να επιλέγουν το σχολείο που θέλουν να πάνε. Όχι μόνο γιατί αυτό είναι σημαντικό να διατηρήσει την, τα κίνητρά τους να μείνουν στο σχολείο, αλλά για να έχουν και ένα ευρύ γνωσιακό πλαίσιο και τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους δώσουν μια θέση εργασία στο μέλλον. Πρέπει να υποστηρίξουμε επίσης και τις μικρές ομάδες διδασκαλίας για τα παιδιά με ειδικά προβλήματα που χρειάζονται περισσότερη προσοχή γιατί αυτό μπορεί να τους βοηθήσει πάρα πολύ και να αποτρέψει την πρόορια κατάληψη. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και βοηθούς εκπαιδευτικούς που επικουρούν τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία και υπάρχουν τέτοιου είδους θέσεις εργασίας σε πολλές χώρες δίνοντας πολύ μεγαλύτερη βοήθεια στους μαθητές που χρειάζονται πιο πολύ χρόνο και πιο πολύ υποστήριξη. Επίσης το να έχουμε <clears throat> υψηλής ποιότητας προσχολική φροντίδα, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ένα θετικό αντίκτυπο και μειώνει το ποσοστό εγκατάλειψης. Η έκθεσή μου έχει συνταχθεί πριν από λίγο καιρό μονάχα και ήταν από τα κύρια πορίσματά μου. Πρέπει να δούμε λοιπόν όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την πρώτη εγκατάλειψη και τα πρώτα χρόνια την προσχολική και πρώιμη σχολική ε, παιδεία είναι ένα συνεχές η παιδεία και δεν μπορούμε να βλέπουμε κατακαιρματισμένα <clears throat> ορισμένες στιγμές τη σχολική πορεία ενός παιδιού γιατί πρέπει να δούμε όλη την πορεία του. Πρέπει να έχουμε περισσότερες σύνδεση και με τους γονείς και με την ευρύτερη κοινότητα. Το είδα αυτό στην προηγούμενη μου έκθεση πόσο σημαντικό είναι. Θα πρέπει λοιπόν να περιλάβουμε αυτή την μέρημνα και για την πρόορη εγκατάλειψη και αυτούς οι οποίοι μένουν στο σχολείο περισσότερα χρόνια. Θα πρέπει οι οργανώσει των νέων, η ΜΚΟ και άλλοι φορείς να εμπλακούν πλήρω σε αυτή την πολιτική και θα πρέπει να σκεφτούμε να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία δικτύων από διάφορα τμήματα της κοινότητα που θα δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα στα άτομα να ξεπεράσουν τα φράγματα που τους εμποδίσουν να έχουν μια καλή παιδεία και φυσικά παίζουν και σημαντικό ρόλο οι γονεί. Ξέρω ότι οι γονεί των παιδιών που έχουν ε, μειονεκτήματα που είναι ανάπηρα δεν εμπλέκονται όσο πρέπει να εμπλέκονται και φυσικά οι αναπηρίε είναι ένας κυριότερος λόγος πρόορη εγκατάλειψη. Επομένως, στο βαθμό του δυνατού θα πρέπει να εμπλακούν και οι γονεί, ώστε να συνεργάζονται με όλους τους άλλους που εμπλέκονται στη σχολική παιδεία. Πρέπει φυσικά να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα των εθνοτικών μειονοτήτων <clears throat> στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης και αυτό είναι ένα κομβικό θέμα και μας επαναφέρει σε αυτά που λέγαμε για, τις, ε, για τους αστικούς πυρήνες. Σε πολλές από τις μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου και σε άλλες μεγάλες πόλεις του, της Ευρώπης υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Η, Δεύτερη ευκαιρία επίση είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα, να ενθαρρύνουμε του μαθητέ οι οποίοι για κάποιο λόγο έχουν εγκαταλείψει το σχολείο να επανέλθουν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο με τον πιο εύκολο δυνατό τρόπο. <clears throat> θα προτιμούσαμε να μην φύγουν από το σχολείο καταρχήν, αλλά μια και φύγανε θα πρέπει να τους δώσουμε μια δυνατότητα να επανέλθουν και να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες τους, να κατανοήσουμε ότι οι μαθητές οι οποίοι απογοητεύτηκαν από την παιδεία μπορεί να δυσκολευτούν να γυρίσουν, αλλά σε μακρόπνο, μακροπρόθεσμο επίπεδο θα είναι για το καλό τους. Επομένως, όχι μόνο αποτροπή της πρόορης εγκατάλειψης, αλλά μας ενδιαφέρει να δίνουμε και δεύτερες ευκαιρίες. Και εν κατακλείδη, χάρηκα που άκουσα ότι τα κράτη-μέλη εξετάζουν το πρόβλημα αυτό και ότι ο στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάλυση και την έρευνα του φαινομένου πρόορης εγκατάλειψης και ελπίζω ότι και το έργο το οποίο κάνουμε και η έκθεσή μου θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου και μας γκαρδιώνει το να βλέπουμε ότι δίνεται μια προτεραιότητα στο θέμα της πρόορης εγκατάλειψης και αντιμετωπίζεται πρεπόντος. Χαίρομαι που θα υπάρχει η ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου που θα κοιτάζει σε κάθε κράτος μέλος τι γίνεται και τις εθνικές στρατηγικές και ελπίζω ότι αυτό θα είναι πραγματικότητα μέχρι το τέλος του 2012. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ για την πρόοδο αυτή και είναι τιμή μου που μπόρεσα να σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση που πιστεύω ότι θα μπορέσει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Ευχαριστούμε κύριε Χάνιμπαλ. Αρχίζει η συζήτηση με τον κύριο Τάκουλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Τρία σημεία. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν την κυρία Χόνεμπολ για την εξαιρετική της εργασία. Και εγώ είμαι ιδιαίτερα ενθουσιώδης με αυτό το θέμα. Και όταν κάποιος είναι ενθουσιώδης ξεπηδίζει πραγματικά τα πράγματα. Και αυτό απαιτεί χρόνο. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Υπάρχει όμως κάτι που θα ήθελα να το δω σε αυτό το κείμενο. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα προς τα κράτη-μέλη, προς τους κυβερνήτες μας. πρέπει καταρχήν να μπορέσουμε να έχουμε συγκρίσιμα μέτρα. Γνωρίζω ότι οι Υπουργοί Παιδείας ήδη το συζήτησαν το θέμα. Εξεπλάγει όταν άκουσα ότι από τη μεριά τους δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στα, συστήματα, στα παιδαγωγικά συστήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα. Όπως πρέπει να τονίσουμε όμως και τα θετικά παραδείγματα. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο πρέπει να έχουμε ένα μέτρο. Να μπορούμε να ταξινομήσουμε έχοντας μια μονάδα μέτρησης. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει στρατηγική για τους δασκάλους. Θα μπορούσαμε ίσως σε αυτό το πλαίσιο να λάβουμε υπόψη μας και αυτό το ειδικό πρόβλημα. Μιλάμε για τη συνεχή κατάρτιση των διδασκόντων. Πολύ ωραία. Αλλά ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την κατάρτιση για να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα. Τρίτο σημείο. Βρισκόμαστε σε περίοδο ισχνών αγελάδων. Καμία χώρα δεν είναι πλούσια εντό εισαγωγικών ή επαρκώ πλούσια. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το εύρος του προβλήματος, την έκταση του προβλήματος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάνουμε οικονομίες στη διδασκαλία αυτό έχει επιπτώσεις. Πρέπει να επιμείνουμε στην ποιότητα της διδασκαλίας και κυρίως στην φάση της προσχολικής ηλικίας. Πρέπει να συνεχίζουμε να επενδύουμε όλο ένα και περισσότερο για να εγγυθούμε ένα καλύτερο μέλλον. ακόμα, ένα, ακόμα ένας εκπρόσωπος από τη Φιλανδία. Λοιπόν, λαμβάνει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και η μελέτη και η έκθεση είναι ιδιαίτερα ποιοτικέ. Ευχαριστώ όλους. Εκτιμώ ιδιαίτερα το σημείο εκείνο όπου αναφέρεται η βοήθεια και η συμβουλή προς τους νέους. Το ακούσαμε και από την μελέτη αλλά και από την εισηγήτρια. Βέβαια από το Συμβούλιο ακόμη δεν ακούσαμε τίποτα τέτοιο. Πρέπει επίσης να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς να ενθαρρύνουμε τους νέους να, να προστρέχουν προς τέτοιες υπηρεσίες Ξέρω ότι στο σχολείο το κοιτάνε οι μαθητές με στραβό μάτι όταν κανείς πάει να τους δώσει καμιά συμβουλή. Πρέπει κατά συνέπεια να τους ενθαρρύνουμε να ζητάνε αυτές τις συμβουλές. Ευχαριστώ. Ο κύριος ο Άνταμ. Σας ευχαριστώ <clears throat> Πρόεδρε και την κυρία Χάνιμπολ θέλω να ευχαριστήσω για την τόσο σημαντική της έκθεση που έρχεται ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Όπως είπαμε, αυτή είναι η αρχή μιας νέας και πιο εντατικής φάσης εργασίας στον τομέα αυτό. Είχαμε πράγματι το στόχο για, την, ε, για το 2010 σε επίπεδο παιδείας, ο οποίος δεν επιτεύχθηκε, γι' αυτό τώρα αναδιατυπώνεται και του δίνεται μεγαλύτερος πολιτικός ρόλος, όπως τόνισαν και όλοι οι ομιλητές. Υπάρχει ένα στοιχείο που θέλω να σας δείξω για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Είναι το θέμα της ανεργίας των νέων που βρίσκεται τώρα στο 20% και ανέρχεται. Η ανεργία για αυτούς που έχουν καταλήψει πρόωρα το σχολείο είναι 50% και αυξάνεται. Αν θέλουμε λοιπόν πραγματικά να επενδύσουμε στην υπερ... υπέρβαση της κρίσης, αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί η δημογραφική αλλαγή είναι εναντίον μας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν όλο το ταλέντο των νέων στη μορφή που μπορεί να το εκφράσει. Από την πλευρά της Κομισιόν θέλουμε να τονίσουμε ότι η προλήψη είναι καλύτερη από την εκ των υστέρων αντιμετώπιση. Όσο ταχύτερα γίνεται αυτή η αντιμετώπιση, τόσο πιο αποτελεσματική προς το, ως προς το κόστος όφελος είναι αυτή η διαδικασία. Η παροχή δεύτερη ευκαιρία είναι σημαντικό παράγον. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε αυτού οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο έχουν βρεθεί εκτό του σχολικού συστήματο. Το σημαντικό στοιχείο λοιπόν είναι η δεύτερη ευκαιρία να τους ξαναοδηγεί στον εκπαιδευτικό κορμό και στην αναγνώριση προσόντων. Και υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες οι οποίες απλώς είναι ένα είδος παρκαρίσματος για άτομα με προβλήματα και δεν τους προσφέρουν καθόλου τα προσόντα που χρειάζονται στην ε, αγορά εργασίας. Η σωστή κατεύθυνση λοιπόν είναι απαραίτητη και είναι κάτι το οποίο δεν πραγματοποιείται πολλές φορές υπέρ των ατόμων που το χρειάζονται περισσότερο. Υπάρχουν και θετικές ε, απολύξεις και αρνητικές. Οι θετικές είναι ότι η πρώτη εγκατάλειψη είναι πάντα, σχεδόν πάντα το τέλος μιας διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει και προειδοποίησεις οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν από τις κατάλληλες πολιτικές. Το βλέπουμε αυτό σε πολλά κράτη-μέλη. Ίσως οι κατοχώρες είναι το καλύτερο παράδειγμα. Βλέπουμε ότι όταν έχουμε μια πραγματικά στοχευμένη πολιτική μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της σχολικής αποχώρησης αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί όπως έχει ληφθεί, λεχθεί προηγουμένως είναι ένα πολυεδρικό πρόβλημα η πρώτη εγκατάλειψη έχει να κάνει με τις οικογένειες, με τις δυσμενείς συνθήκες, έχει επιπτώσεις σε επίπεδο εργασίας κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού πάρα πολύ εμπλεκόμενοι και αυτό φυσικά έχει διαφορετική μορφή σε κάθε χώρα κάθε χώρα έχει διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικά προβλήματα πρόορης εγκατάλειψης. Ναι. Τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να έχουν εθνικές στρατηγικές, πρέπει όμως να είναι αρκετά εύκαμπτες και αρκετά στοχευμένες αυτές οι στρατηγικές για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα επίπεδα και όλα αυτά τα αίτια που προκαλούν την σχολική εγκατάλειψη. Άρα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για συλλογή στοιχείων. Πολύ λίγες χώρες αυτή τη στιγμή <clears throat> καταγράφουν πλήρως και αναλύουν τους λόγους για τη σχολική εγκατάληψη και την, ε, τον επιπολασμό του φαινομένου κατά περιοχή και κατά ομάδα του πληθυσμού. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια σωστή αντιμετώπιση πρόληψης και αντιμετώπισης παροχής δεύτερης ευκαιρίας όπως θέλετε να το διατυπώσετε και μέτρα πρόληψης και μέτρα επανενσωμάτωσης. Αν λοιπόν όλα αυτά συντονιστούν σωστά, θα πρέπει συγχρόνως να ανταποκρίνονται και στις ιδιαίτερες συνθήκες. Επομένως, σε εθνικό επίπεδο χρειάζεται και στοχοθεσία και ευκαμψία, ώστε το μείγμα αυτό να είναι πράγματι αποτελεσματικό. Και εδώ μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει κάποιο ρόλο, μπορεί η έκθεση του Κοινοβουλίου να είναι χρήσιμη και όπου το έργο της Κομισιόν μπορεί να δώσει υποστέμενη αξία σε τρεις συγκεκριμένους τομείς. Πρώτον, με την ανοιχτή μέθοδο συνεργασίας, γιατί σχεδόν όλα αυτά τα μέτρα για τα οποία μιλάμε είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. τα κράτη-μέλη όμως έχουν πολλά να μάθουν από την εμπειρία των άλλων κρατών μελών Υπήρξε στο παρελθόν συνεργασία επί τη βάση της ανοιχτής μεθόδου συνεργασίας για την ανοιχτή μάθηση και τα προβλήματα κοινωνικού χαρακτήρα αλλά και την πρόορη εγκατάλειψη και το φθινόπωρο θα δημιουργήσουμε και μια νέα ομάδα υψηλού επίπεδου με εκπροσώπους των κρατών μελών για να παρακολουθήσει την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών όπως αναφέρονται στη σύσταση. Πιστεύω λοιπόν και η έκθεση του Κοινοβουλίου θα παίξει κάποιο ρόλο για αυτά. Θα ξεκινήσουμε μελέτες με δική μας πρωτοβουλία μέσα στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα για να έχουμε περισσότερα στοιχεία, να ξέρουμε ποιες πολιτικές είναι εύστοχες και μπορούν να θεωρηθούν πρόσφορες για την αντιμετώπιση του προβλήματος και μπορούμε να επαναλάβουμε και τη συνδιάσκεψη που έγινε πέρσι σε σχέση με τη σύνδεση σχολείου και επιχειρήσεων, όπου τονίστηκαν πάρα πολλά τέτοια θέματα που αναφέρθηκαν και σήμερα, ότι η συμμετοχή και παραγόντων από τις τοπικές επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά που δεν θεωρούν ότι αξίζει το σχολείο, αλλά αν δουλεύουν με τις τοπικές επιχειρήσεις και τους βλέπουν έρχονται στα σχολεία και τους παρέχουν μια νέα μορφή, διαφορετική μορφή κατάρτισης, μπορεί να τους ενδιαφέρει περισσότερο. Μπορούμε να βοηθήσουμε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βέλτιστες πρακτικές που παρουσιάζονται σε συνδιασκέψεις που μπορούν να βοηθήσουν. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προσθέσουμε προσθέμενη αξία. Ο δεύτερος είναι με το πρόγραμμα διαβίου μάθησης και τους διαδόχους του. Έχουμε πολλά θετικά σχέδια που λαμβάνουν χώρα, ιδίως μεταξύ του κομμένου Εταιρικές Σχέσεις και κομμένου Ρέτζιο, και βασίζεται τα προγράμματα αυτά σε αντιμε... ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ περιοχών και σχολείων. Είναι λοιπόν από τις πρωτοβουλίες που δουλεύουν σε επίπεδο βάσης και ευνοούν και τους διδάσκοντες και τους μαθητές που μπορούν να μεταλαμβαδεύσουν την εμπειρία τους και να διδάξουν εαυτούς και αλλήλους. Δεν είναι λοιπόν μια εκ των άνω επιβολή λύσεων, αλλά είναι η καινοτομία σε επίπεδο βάσης. Θα είναι πάρα πολύ θετικό λοιπόν αυτό. Και επίσης για τα διαφορετικά ταμεία που είναι η κυριότερη πηγή χρηματοδότησης για τις υποδομές και την εκπαίδευση και τις πρωτοβουλίες μέσα στα κράτη-μέλη έχουν τεράστιο δυναμικό το οποίο υποαπασχολείται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα έκθεση κάπως ανησυχητική από το Ελεκτικό Συνέδριο το 2006 που βλέπει το πώς οι διαθωτικοί πόροι έχουν <clears throat> μειώσει την πρόορη εγκατάλειψη. Βρήκαν ότι υπήρχε κάποιος αντίκτυπος, αλλά ήταν πολύ περιορισμένη η αποδοτικότητα, γιατί δεν υπήρχε η σωστή μορφή συντονισμού και η απαραίτητη συνοχή των πρωτοβουλειών αυτών μεταξύ των κρατών μελών. Γι' αυτό χρειάζεται μια πιο στρατηγική προσέγγιση στη χρήση των διαθωτικών πόρων στις εθνικές στρατηγικές. Στη νέα φάση λοιπόν είναι ο καλύτερος τρόπος να κάνουμε πιο αποτελεσματική τη λειτουργία των διαφορετικών πόρων για να είναι πιο συνακτική και να ακολουθεί αυτή τη σύσταση. Αυτό είναι λοιπόν το μέλλον για μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Κοινοβούλιο για την έκθεση αυτή που είναι εν εξελίξη και για τη μελέτη που περιμένουμε να λάβουμε σε Περισσότερα λεπτομέρεια. Ευχαριστώ. Thank you very much, Adam. Ευχαριστώ, Άνταμ. Επιθυμεί άλλος κανείς. Εσείς κυρία μου. Όχι. Δεν επιθυμείτε να παρέμβετε. Καλά λοιπόν. Ευχαριστούμε κυρία Χάνιμπολ για τις τροπολογίες προβλέπεται ως ε, προθεσμία η 7η Ιουλίου το μεσημέρι στις 12. Και θα προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι η έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών υπενθυμίζω ότι έχουμε καταργήσει τη συνεδρίαση του τέλους Αυγούστου. Λοιπόν, λάβετε το υπόψη σας και διαγράψετε το από την ε, ατζέντα σας. Υπάρχει καμία ένσταση? Πάει λοιπόν το 9. Επανέρχομαι όμως στο 8, διότι μόλις ο γραμματέας με διορθώνει. Η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών είναι η 6η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη. 6η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη. Το 10 που είναι τα διάφορα. Δεν βλέπω κανείς να έχει κανένα διάφορο.